Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίσατε να καλωσορίσουμε και τους βουλευτές, τους βοηθούς και όποιον θέλει να συμμετέχει και να καλωσορίσω και τα μέλη της Επιτροπής ΕΜΒΗ γιατί αυτή η ακρόαση θα γίνει από κοινού. Ε, έχουμε τις δύο ε, επιτροπές. Ε, καλωσορίζω λοιπόν και τον συνάδελφο από την Επιτροπή ΕΜΒΗ. Ε, προφανώς και μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τι ε, θα ε, μας πούν οι εμπειρογνώμονες για την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη και τα όσα μας περιμένουν στο μέλλον. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνδιοργανώνει αυτή την ακρόαση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη, την οποία αποκαλούμε ELD, ε, τέθηκε σε ισχύ Στι 30 Απριλίου του 2004, τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν τρία χρόνια για να μεταφέρουν την οδηγία στο εσωτερικό τους ε, δίκαιο και η μεταφορά της ε, ELD ολοκληρώθηκε τελικά τον Ιούλιο του 2010. Πάνω από τρία χρόνια, αλλά τέλο πάντων τα καταφέραμε. Βάσει του άρθρου 18 τη οδηγία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε το 2014 να εκπονήσει έκθεση για την εμπειρία από την εφαρμογή της οδηγίας στην πράξη και βεβαίως έχουμε και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς εφαρμόστηκε αυτή η οδηγία επί τη βάση και των εθνικών εκθέσεων που καταρτίστηκαν το 2013 από τα κράτη-μέλη και υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλων σχετικών πληροφοριών. Λόγω των καθυστερήσεων ε, στις εκθέσεις ε, και στην αξιολόγηση, αλλά και λόγω και των αλλαγών που έγιναν σε πολιτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014, η έκθεση εγκρίθηκε τελικά τον Απρίλιο του 2016. Πλέον ολοκληρώθηκε ο κύκλος και θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την ακρόαση η οποία θα είναι λίγο πιο συγκεκριμένη επί των σημείων αυτών και θα μπορέσουμε να έχουμε και κάποιες πληροφορίες. Οι επιτροπές ε, Γιούρι και Έμβη είναι οι αρμόδιες ε, επιτροπές για την έγκριση της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη και θεωρήσαμε λοιπόν ότι... Ε, τα μέλη της Επιτροπής άλλωστε είπαν ότι το σωστό θα ήταν οι δύο επιτροπές ε, να είναι αρμόδιες και πάλι όσον αφορά την επόμενη έκθεση εκτέλεσης. Και κατά συνέπεια λοιπόν έχουμε αυτή την ακρόαση η οποία συνδιοργανώνεται από τις δύο επιτροπές ε, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό που μας ενδιαφέρει όπως αναφε... καταλάβατε πολύ καλά. Σήμερα λοιπόν έχουμε κάποιους εμπειρογνώμονες, ε, ομιλητές και εκπροσώπους ε, διαφόρων συμφερόντων, καθώς επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη ε, επεξεργασία των συνεπειών της ε, μεταφοράς της οδηγίας αυτής για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις και για το περιβάλλον και οτιδήποτε άλλο θα έλεγα το οποίο θα μπορούσε να ε, ληφθεί υπόψη και θεωρείται απαραίτητο για, τη για την οδηγία αυτή. Χωρίς να καθυστερήσω περαιτέρω να δώσω το λόγο στον το ομιλητή, αν μου επιτρέπετε κυρία Ζαβόρ, πρόκειται για την κυρία Σάντρα Κασότα από το Παρεπιστήμιο της και για να μας μιλήσει για τις ε, συγκεκριμένες πτυχές της μεταφοράς της οδηγίας, πιο συγκεκριμένα το κατόφλι σημασίας δηλαδή ε, το μέγεθος της περιβαλλοντικής ευθύνης, καθώς επίσης και τις εξαιρέσεις ε, και τις παρεκκλήσεις που προβλέπονται. Με την άδειά σας λοιπόν ε, να ακούσουμε την πρώτη ομιλήτρια. Παρακαλώ κυρία μου έχετε το λόγο. Για ένα τέταρτο και από εκεί και πέρα για να διευκολύνουμε και τις εργασίες και για να μην καθόμαστε να σας παρακολουθούμε εγώ και ο κύριος Ζαβόρ, έχετε ρολόγια στις οθόνες, οπότε μπορείτε να παρακολουθήσετε αν είστε μέσα στο χρόνο. Κυρίες και κύριοι, είναι τιμή μου που με προσκαλέσατε σήμερα να μιλήσω για την οδηγία για την ε, περιβαλλοντική ευθύνη. Τα κράτη-μέλη είχαν μέχρι το 2007 προθεσμία για να προωθήσουν ε, και να μεταφέρουν αυτή την οδηγία και τώρα μπορούμε να αξιολογήσουμε τη διαδικασία της εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η οδηγία αυτή είναι αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας ε, πάνω από 8 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελέτησε και συζήτησε την έννοια του νομοθετικού ε, πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθόρισε και τα βασικά κριτήρια για ε, τα περιβαλλοντικά θέματα και τις περιβαλλοντικές ευθύνες. Το κείμενο της οδηγίας λοιπόν είναι αποτέλεσμα διαφόρων συμβιβασμών σε πολιτικό επίπεδο και το κείμενο της οδηγίας είναι πάρα πολύ διπλωματικό. Σας διακόπτω, μου λένε ότι δεν υπάρχει διερμηνία από τα γαλλικά. Μήπως θα μπορούσατε να διορθώσετε αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε. Έλεγα λοιπόν ότι το κείμενο της οδηγίας είναι πάρα πολύ διπλωματικό κείμενο. Δεν ε, αναφέρεται ρητά σε κάτι συγκεκριμένο, ούτε καν στα πολύ βασικά στοιχεία της, του νέου καθεστώτος περιβαλλοντικής ευθύνης του οποίο θέλησε να συμπεριλάβει. Όπως για παράδειγμα τη αυστηρά θέματα ευθύνης. Ε, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι αυτά που βλέπετε εδώ στη διαφάνεια, στις οθόνες, είναι ε, σημεία τα οποία είναι κοινά σε όλα τα επίπεδα νομοθεσίας, είτε πρόκειται για περιφερειακά, διεθνή ε, νομοθεσία των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν είναι τυχαία η σειρά ε, με την οποία ιεραρχούνται. Ακολουθούν μία ε, λογική ακολουθία και επομένως εάν το πρώτο σημείο που είναι ο ορισμός της περιβαλλοντικής ζημίας αλλάξει, τότε αυτό θα έχει συνέπειες και σε όλα τα υπόλοιπα σημεία. Να περάσω λοιπόν κατευθείαν στο προκείμενο και να σας πω ότι για το πρώτο σημείο, το οποίο είναι ο ορισμός της περιβαλλοντικής ζημίας και το κατόφλι ε, από το οποίο ξεκινά θα πρέπει να αλλάξει. Διότι εάν αλλάξει ο ορισμός, αυτό θα ε, αντανακλάται και σε όλα τα υπόλοιπα σημεία. Η σημερινή μου παρέμβαση θα επικεντρωθεί σε τρία βασικά σημεία Πρώτον, ε, τον ορισμό της περιβαλλοντικής ζημίας και την έννοια του κατοφλίου. Δεύτερον, το πεδίο εφαρμογής και τρίτον, τις παρεκκλήσεις. Όταν λοιπόν μπορεί ο υπεύθυνο να αποφύγει την ευθύνη επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες παρεκκλήσει. Ο ορισμός της περιβαλλοντικής ζημίας είναι αρκετά περιοριστικός ω έννοια. Πρόκειται για έναν ορισμό ο οποίος περιλαμβάνει ε, τρεις ε, κατηγορίες συγκεκριμένων φυσικών πόρων, ζημία σε προστατευόμενα είδη και σε φυσικούς σκοτόπους, ε, όπως ορίζεται από την οδηγία Habitat και για τα λεπτά, η, οδηγία, η ζημία προς τα ύδατα όπως ε, καθορίζεται από την οδηγία στα ύδατα και η ζημία στη γη όπως καθορίζεται από τη ρήπανση του εδάφους. Και αυτό φυσικά ε, έχει και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Εδώ λοιπόν η νομοθεσία είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται ε, ως ε, ε, αναφορά παραπομπή ο νομοθέτης αποφασίζει να ορίσει την έννοια της περιβαλλοντικής ζημίας ε, αναφερόμενος παραπέμποντας σε άλλες οδηγίες και ο ορισμός δεν περιλαμβάνει και την συνήθη ζημία που είναι ζημία αγαθών και προς τρίτους. Έχουμε λοιπόν περιβαλλοντική ζημία φυσικών πόρων τα οποία ακολουθούν ένα οικολογικό όραμα και όχι ανθρωποκεντρικό όραμα. E uh, Ο Ευρωπαίος νομοθέτης λοιπόν επέλεξε να συμπεριλάβει στο κείμενο για να ορίσει την περιβαλλοντική ε, ζημία έναν τεχνικό ορισμό αλλά δεν έχει ένα μη τεχνικό νομικό ορισμό. Πρόκειται για έναν επιστημονικό τεχνικό ορισμό, αλλά δεν είναι τεχνικός από νομική σκοπιάς, διότι αν εξετάσουμε το άρθρο 2 του ορισμού που βλέπετε εδώ στη διαφάνεια λέει ότι η περιβαλλοντική ζημία σημαίνει μετρήσιμη αλλαγή σε φυσικούς πόρους ή μετρήσιμη παρακόλληση φυσικών πόρων που μπορεί να προκύψει άμεσα ή έμεσα. Άρα πρόκειται για επιστημονική ορολογία η οποία δεν έχει συγκεκριμένα και σαφή κριτήρια. Επιτρέπει να δοθούν διάφορες ερμηνείες από τα κράτη-μέλη σε διάφορα εθνικά συστήματα. To have a, definition that can fix... Και ε, πρέπει να έχουμε έναν ορισμό ο οποίος θα πρέπει να θέτει έναν ελάχιστο κοινό παρανομαστή ο οποίος όμως ο ορισμός θα είναι νομικός και όχι επιστημονικός, διότι αν μείνει ως έχει, ε, να έχουμε δηλαδή έναν επιστημονικό κοινό παρανομαστή τότε ο δικαστής θα αντιμετωπίζει δυσκολίες και δεν θα μπορεί να τον κατανοήσει. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ έγκυται στο γεγονός ότι ο επιστημονικός ορισμός επιβάλλει πολύ υψηλό ε, όριο από το οποίο θεωρούμε ότι υπάρχει περιβαλλοντική ζημία και το όριο το οποίο επιβάλλεται είναι τόσο υψηλό το οποίο είναι αδύνατο να το υπερβούμε σε αρκετές περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποια μορφή ζημία. Υπάρχει λοιπόν κατά την άποψή μου ε, πολύ επιστημονική ορολογία χωρίς να υπάρχει κάποια κοινή δράση στον ορισμό της περιβαλλοντικής ζημίας που θα μπορούσε να γίνει κατανοητή, να την αντιληφθούν και να την εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Ε, πρέπει να υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα όρια και ακριβή κριτήρια για να μπορέσουμε το, ε, να έχουμε έναν μηχανισμό ευθύνη ο οποίος να είναι αποτελεσματικός ε, και να, μετα... να είναι αποτελεσματικός είναι το χρόνο. διότι ο μηχανισμός της ευθύνης αυτή τη στιγμή δεν είναι λειτουργικός. Το δεύτερο σημείο ε, είναι το πεδίο εφαρμογής, ε, το δεύτερο σημείο που μας ενδιαφέρει. Δεν έχω και πολλά να σας πω εδώ, διότι το πεδίο εφαρμογής εξαρτάται σε πολύ αυστηρό βαθμό από τον ορισμό της περιβαλλοντικής ζημίας. Στον ορισμό λοιπόν τον οποίο ε, ε, επέλεξε οι κατόπιν διαπραγμάτευση. διότι το πεδίο εφαρμογής ε, στην πραγματικότητα είναι λογική συνέπεια. Ο ορισμό και το πεδίο εφαρμογή είναι οι δύο πλευρέ του ιδίου νομίσματος. Είναι πάρα πολύ περιοριστικό λοιπόν το πεδίο εφαρμογή γιατί οι δραστηριότητε οι οποίες υποσκάπτουν την περιβαλλοντική ζημία περιλαμβάνονται στο παράρτημα 3, που καθορίζουν τον πιθανό δυνητικό κίνδυνο προ την υγεία και το περιβάλλον. Ε, ο κατάλογος της οδηγίας αναφέρει επίσης ε, και τους ε, προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτές τις δραστηριότητες, παραδείγματο χάρη πρώτερη έγκριση, ειδικέ προϋποθέσεις, καταχώρηση κλπ. Αλλά σε αλλαγές ή ζημία στην βιοποικιλότητα η μέθοδος επιλογής και η επιλογή της επαγγελματικής δραστηριότητας δεν εφαρμόζεται, διότι η ευθύνη επεκτείνεται σε κάθε πιθανή δραστηριότητα, αρκεί να μπορούμε να αποδείξουμε ευθύνη ή αμέλεια. Η πετιότητα μάλλον ή αμέλεια. Και αυτό φυσικά σημαίνει ότι έχουμε μια τεκτική επέκταση ή διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή, διότι επιτρέπεται ε, στα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη του και κάποιε άλλε δραστηριότητε πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 σε περίπτωση αμέλεια και αυτό είναι αρνητική συνέπεια και αυτή η εθελοντική επέκταση σημαίνει ότι θα αυξήσει και τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Διότι κάποιες αρμόδιες αρχές θα πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα από άλλες. Και αυτό φυσικά θα αυξήσει την έλλειψη ισορροπίας και εναρμόνισης. Τώρα, το τελευταίο σημείο στο οποίο θα επικεντρωθούμε είναι οι εξαιρέσεις, οι παρεκκλήσεις. Αυτός ε, είναι όταν οι περιπτώσεις στις οποίες ε, ο υπεύθυνο ε, αποφεύγει την ευθύνη, δεν θεωρείται υπεύθυνο και έχουμε δύο μορφές παρεκκλήσεων. Έχουμε εξαιρέσεις και... και άμυνες. Αν δείτε το άρθρο 4 εδώ στις διαφάνειες, θα δείτε ότι εξαιρέται ευθύνη ζημία λόγω κλιματικής αλλαγής. Όταν είναι αδύνατον να καθορίσουμε ε, η πετιότητα που είναι η σχέση μεταξύ της ζημίας και του γεγονότος. Ε, αν έχουμε για παράδειγμα οξύνη ή ε, ρήπανση, περιπτώσεις τις οποίες δεν μπορούμε να έχουμε πετιότητα. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις εξαιρέσεων για την ε, περίπτωση ανωτέρας βίας, ε, ένοπλη σύραξη, εμφύλιος πόλεμος. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει ευθύνη του ε, ε παραγωγού ή του φορέα και σε αυτή την περίπτωση η εξαίρεση είναι υποχρεωτική. Επίσης έχουμε εξαιρέσει σε περίπτωση πετρελοκυλίδας, πυρηνικής καταστροφής, αρκεί να καλύπτονται από διεθνείς συμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν ένα παράρτημα 4 αλλά θα πρέπει να σας πω εδώ ότι όλες αυτές οι συμβάσεις ε, στην πραγματικότητα δεν ε, είναι αποτελεσματικές. Επομένως, Έχουμε μια δεύτερη κατηγορία εξαιρέσεων, ε, τις αμυντικές περιπτώσεις, είναι οι προαιρετικές, οι οποίες δεν ισχύουν διαβίου και έχουμε δύο περιπτώσεις λόγω άδεια και λόγω εξέλιξη της τεχνολογίας. Ε, Επομένω, είναι οι περιπτώσει ε, λόγω άδεια όπου μια εθνική αρχή ή κράτος μέλος ε, παράγει κάποιο προϊόν ή εκπέμπει κάποιες ουσίες. Για παράδειγμα, φορέα, ο οποίος ε, ε, εκμεταλλεύεται απόβλητα, ο οποίος είναι κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων λόγω ε, ρητή άδεια από τις αρχές ή από το κράτος μέλος. Και έχουμε και την, τα αμυντικά επιχειρήματα λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας. Όταν δεν είναι κάποιο φορέας υπεύθυνο, διότι χρησιμοποιεί ένα προϊόν το οποίο όταν ε, διέθεσε το προϊόν στην αγορά δεν είχε αποδειχθεί ότι θα μπορούσε να έχει επιζήμιες συνέπειες ε, λόγω των ε, επιστημονικών γνώσεων που είχαμε για παράδειγμα. Σκεφτείτε για παράδειγμα τους παραγωγούς γενετικών τροποποιημένων προϊόντων και αυτών που χρησιμοποιούν νανοτεχνολογίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις το πρόβλημα ε, της οδηγίας είναι ότι δεν βασίζεται στην ε, μετατόπιση του βάρους της απόδειξης και δεν συνδέει την αυστηρή ευθύνη με τη μετατόπιση του βάρους της απόδειξης. Άρα αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη έχουν πολύ μεγάλη ελευθερία ε, ελευθερία κινήσεων και ουσιαστικά τα κράτη-μέλη θα χρησιμοποιήσουν την ευθύνη και όχι την αυστηρή ευθύνη, γιατί η ευθύνη λόγω υπετιότητας είναι πάρα πολύ δαπανηρή. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι δεν ε, είναι πολύ θετική η οδηγία. Όπως θα δείτε στις διαφάνειες αυτές, προσπάθησα να καταλάβω την αναλλαγία. Γιατί ο Ευρωπαίος νομοθέτης ήθελε αυτές τις αναλλαγίες. Υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσει. Η ισότητα και η ισορροπία. Η ισότητα γιατί δεν είναι δίκαιο να υποχρεώνεται ένας παραγωγός ε, να πληρώνει ε, για κάτι το οποίο δεν γνώριζε τότε ε, κατά την άσκηση της δραστηριότητας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζημία, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να τα σταματήσουμε όλα αυτά, γιατί δεν υπάρχουν και κίνητρα για να σταματήσουν πιθανώς ρηπογόνε δραστηριότητε. Και τίθεται και θέμα ισορροπίας εδώ που είναι και το αιώνιο δίλημα μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης αφενός και από την άλλη προστασίας του περιβάλλοντος. Ε, τα αμυντικά επιχειρήματα στην πραγματικότητα λοιπόν επιτρέπουν πάρα πολλές ε, εξαιρέσεις, έχουν ε, πολύ μεγάλη ελευθερία τα κράτη-μέλη και ε, στην πραγματικότητα ο λόγος ύπαρξης αυτών των ε, ε, αμυντικών επιχειρημάτων είναι παράδοξος. Αν σκεφτεί κανείς ότι συμπεριλαμβάνονται σε ένα κανόνα ο οποίος στόχο έχει να εφαρμόσει την αρχή του ορυπαίνων πληρώνει. άρα στην πραγματικότητα παρακολύω την εφαρμογή διότι στην πραγματικότητα δεν θα πρέπει να είναι άμυρος ευθυνών όποιος ε, δημιουργεί, προκαλεί ζημία, ακόμα και αν δεν υπάρχει υπετιότητα, θα πρέπει κάπως ε, να μπορεί να αποζημιωθεί όλη αυτή η ρήπανση. Και επίσης ε, θα πρέπει να καλύπτονται Cedar, this kind of damage. και η, ο κίνδυνος ανάπτυξης, ζημία που προκαλείται από αυτές τις περιπτώσεις. Όταν για παράδειγμα κάποιος είναι υπεύθυνο στις περιπτώσεις που υπάρχει μια δραστηριότητα που ελοχεύει ο κίνδυνος να είναι ρηπογόνος ή μπορεί να υπάρξει εξέλιξη της ρηπογόνου συνέπειας, δηλαδή ο κίνδυνος εξέλιξης της ρήπανσης. Και στην πραγματικότητα εδώ ε, η οδηγία δεν το λαμβάνει υπόψη της, ενώ περιλαμβάνεται στο γερματικό δίκαιο ως ε, μια συγκεκριμένη ορολογία Entwicklung Risiko στο οποίο μπορούμε να το συμπεριλάβουμε ίσως στην οδηγία. Πλησιάζω τώρα τα συμπεράσματά μου. Όσον αφορά λοιπόν ε, τα κατόφλια, ε, που είναι το πρώτο θέμα που μου ζητήθηκε να σας ε, αναφέρω, η έννοια της ε, περιβαλλοντικής ζημίας θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ελάχιστο κατόφλι, το οποίο θα πρέπει από εκεί και πέρα να λειτουργεί κλιμακότα και δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από τα κράτη-μέλη, αλλά και από περιφέρειες ή από τοπικές διοικήσεις. Θα πρέπει αυτή η κλιματοκοτή εφαρμογή να γίνεται ανάλογα με τις διάφορες χρήσεις και με τα διάφορα μέσα επίσης. Άρα η κλιμακωτή αυτή μέθοδος ε, θα πρέπει να επιτρέπει την εφαρμογή και της αρχής ε, ορυπαίνων πληρώνει, της αρχής επικορικότητας και επίσης και τη συμμετοχή των μη επισήμων φορέων που είναι πάρα πολύ σημαντική για την εφαρμογή της οδηγία. Δεύτερον, το πεδίο εφαρμογής. Το πεδίο εφαρμογής ε, στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ περιορισμένο και θα πρέπει να διευρυνθεί και τέλος, όσον αφορά τις εξαιρέσεις και τα επενδυτικά επιχειρήματα, θεωρώ ότι αποδυναμώνουν το καθεστώς ε, της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη, διότι στην πραγματικότητα αμβλύνουν τις ε, αποκλίσεις ε, και αποφεύγεται η πετιότητα και η πληρωμή ευθυνών. Επιτρέπουν λοιπόν πολύ μεγάλο περιθώριο λιγμών στα κράτη-μέλη, τα οποία αποφασίζουν κατά πόσον θα τις χρησιμοποιήσουν ή όχι και επομένως αντί να ενισχύουν την εναρμόνιση, έχουμε την ε, διόγκωση των διαφορών στην εθνική νομοθεσία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε για την ανάλυση σας και τις εξηγήσεις σας. Ε, δυστυχώς, μόνο δύο λεπτά μας καθυστερήσατε, οπότε άξιζε το κόπο. Και τώρα... Ε, ο λόγος στον Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΜΒΗ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές που είναι εδώ. Θα ήθελα να δώσω αμέσως το λόγο στον επόμενο ομιλητή, τον Dr. Crystal Smith από το Πανεπιστήμιο του Μάστριχ, το οποίο θα μιλήσει για την ε, σημασία των, ε, της ασφάλειας και των φορέων λειτουργίας για την κατάσταση σε ένα περιβάλλον ε, ανταγωνιστικό και κάποια μορφή ειδικών ταμείων. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Η καθηγήτρια λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να σας παρουσιάσω τις απόψεις μου για την υποχρεωτική οικονομική ασφάλεια. Δεν θα ήμουν ακαδημαϊκός αν δεν ξεκινούσαμε λίγη θεωρία. Εξέτασα λοιπόν ε, την ε, οδηγία για την ε, περιβαλλοντική ευθύνη από άποψη νομική και οικονομική που εξετάζει πώς το κάθε άτομο αντιδρά στις αλλαγές στην νομοθεσία και υπό ποιες συνθήκες ένας κανόνας μεγιστοποιεί την κοινωνική ευημερία. Ο περιβαλλον, Η περιβαλλοντική νομοθεσία λοιπόν έχει ως στόχο μία δραστηριότητα ενός εφορεία διαχείρισης ή λειτουργίας ε, που μπορεί να κοινωνικά ε, να είναι υποφελής να βλάπτει το περιβάλλον, αλλά ο Ριπένον δεν λαμβάνει το περιβάλλον ως ε, υπόψη του, διότι το θεωρεί εξωτερικό παράγοντα. Έτσι λοιπόν μειώνει την κοινωνική ευημερία. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε το δίκαιο των αδικοπραξιών για να μπορέσουμε να αναγκάσουμε τον operator να πάρει υπόψη του αυτό το εξωτερικό, αυτόν τον εξωτερικό παράγοντα και να φροντίζει το περιβάλλον. Υπάρχουν διάφορες ε, κατηγορίες για να το επιτύχουμε αυτό. Είναι το θέμα της αμέλειας και της αντικειμενικής ευθύνης. Υπάρχει ε, προτίμηση για, για την αντικειμενική ευθύνη όταν έχουμε επικίνδυνες δραστηριότητες ε, που βλάπτουν το περιβάλλον και με το επόμενο σχήμα θα σας εξηγήσω το λόγο. Ο κανόνας ε, της αμέλειας δίνει στον φορέα τα κίνητρα να έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο δέουσας επιμέλειας. Πρέπει λοιπόν το δικαστήριο να θεσπίσει ποιο είναι το επίπεδο ε, επιμέλειας και φροντίδας και αν το πληρεί θα εξαιρείται από την ευθύνη. Επί της αρχής λοιπόν, επειδή ο φορέας θέλει να αποφύγει την ευθύνη, θα πάρει κάποιες προφυλάξεις. Προφυλάξεις ως το επίπεδο που θα τον ε, προστατεύει που θα προστατεύεται από οποιαδήποτε ευθύνη. Αν μπορέσει λοιπόν το δικαστήριο να βρει το βέλτιστο επίπεδο, θα είναι εντάξει, αλλά συνήθως είναι δύσκολο. Ο κανόνας της αντικειμενικής ευθύνης τώρα. Σύμφωνα με αυτόν υπάρχει ευθύνη ανεξαρτήτως ε, φροντίδας που έχει ληφθεί. Άρα θα ληφθούν μέτρα μέχρι ένα συγκεκριμένο επίπεδο προφύλαξης και θα σταματήσει να λαμβάνει προληπτικά μέτρα αν τελικά το κόστος είναι μεγαλύτερο από τα ωφέλη. Και στις δύο λοιπόν περιπτώσεις μπορούμε να έχουμε τη αβέλτιστα μέτρα προφύλαξης, όμως για τις επικίνδυνες δραστηριότητες υπάρχει το επιχείρημα ότι είναι πολύ σημαντικό ο δυνητικός ε, μολύνων, ο φορέας, να λαμβάνει μέτρα ε, που ε, ακόμα όλα τα μέτρα, ακόμα και αυτά που δεν θα παρατηρούσε κανείς, είναι το επίπεδο της δραστηριότητας, και για, όπως το ονομάζουμε, και γι' αυτό χρειαζόμαστε την αντικειμενική ευθύνη. Και υπάρχει και το επίπεδο της αφαιρεγγιότητας. Δεν αρκεί η αντικειμενική ευθύνη αν έχει κίνδυνο αφαιρεγγιότητας. Αν ένας ε, φορέας ξέρει εκ των προτέρων ότι αν προκαλέσει περιβαλλοντική ζημία τόσο μεγάλη ώστε να μην μπορεί να την καλύψει οικονομικά, θα είναι αφαιρέγγιος και έτσι δεν θα έχει πλέον κίνητρο για να λάβει τις βέλτιστες προφυλάξεις. Γι' αυτό από θεωρητική άποψη η αντικειμενική ευθύνη δεν θα πρέπει να εισηχθεί με τέτοιες οικονομικές εγγυήσει όπως η αφαιρεγγιότητα γιατί αλλιώς δεν θα διασφαλίσουμε την προστασία από την περιβαλλοντική ζημία. Επίσης θα καταστρέψει την προληπτική δράση της οδηγίας γιατί αν ξέρεις εκ των προτέρων ότι δεν μπορείς να πληρώσεις μια ζημία γιατί να φροντίσεις για αυτήν. Φυσικά είναι ωραία να μιλάμε στη θεωρία. Οι θεωρητικές ιδέες είναι εντάξει, αλλά η πρακτική μπορεί να είναι πιο δύσκολη. Το 2014, όταν συμφωνήθηκε η οδηγία, οι απόψεις ήταν ε, δίσταντος προς τις ε, οικονομικές ε, εξασφαλίσεις. Υπήρχαν ε, λοιπόν διάφορες απόψεις μεταξύ των κρατών μελών και υπήρχαν και αντιθέσεις στην επίπεδο της Κομισιόν. Οπότε έμεινε το θέμα στα κράτη-μέλη. Επίσης, δεν υπήρχε αγορά για εξασφαλίσεις για την περιβαλλοντική ζημία. Πώς να υποχρεώσεις κάποιον λοιπόν να τις έχει. Άρα καταλήξαμε σε μια μετριοπαθή λύση. Άρθρο 14. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πάρουν μέτρα ώστε να καταστήσουν ικανούς ε, τους ε, φορείς ε, να λάβουν τις εξασφαλίσεις εκείνες τις οικονομικές που θα καλύπτουν τους κινδύνους. Θα... Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα κομμάτι ενθάρρυνσης που απαιτείται. Προφανώς λοιπόν τα κράτη-μέλη ακολούθησαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ξεκίνησαν με πληροφόρηση και οδηγήθηκαν σε ένα άλλο επίπεδο όπου θέσπισαν υποχρεωτικά ας πούμε συστήματα για τις οικονομικές εγγυήσεις αλλά ε, προχώρησαν σε μια επιλεκτική ένα επιλεκτικό καθεστώς. Ε, αυτά που είχαν υποχρεωτική την ε, εξασφάλιση έθεσαν κάποια όρια, επίσης συγκεκριμένα ποσά, κατόφλια και ταβάνια και σε κάποιες περιπτώσεις έγιναν και συγκεκριμένες εξαιρέξεις. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει μία ευρωπαϊκή λύση που να θεωρείται η πιο αποτελεσματική. Ήδη δύο φορές η Κομισιόν ε, εξέτασε το κατά πόσο θα έπρεπε να έχουμε μια εναρμονισμένη οικονομική εξασφάλιση σε υποχρεωτικό επίπεδο το 2016 με το REFIT ε, ήταν η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά ήταν το 2010. Στην αξιολόγηση Refit η Κομισιόν είπε ότι αν έχουμε ένα ε, εναρμονισμένο ε, σύστημα οικονομικών εξασφαλίσεων, το εργαλείο αυτό θα παραμείνει ασθενέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι υπάρχει διαφορά στον τρόπο που έχει αναπτυχθεί η ασφαλιστική αγορά στην Ευρώπη. Καλό θα ήταν λοιπόν να υπάρχει σε εθνικό επίπεδο μια εξατομικευμένη λύση. Από την άλλη βέβαια υπήρχε το πρόβλημα των ε, μεγάλη κλίμακας ε, ατυχημάτων και των αφαιρέγγιων φορέων. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της απλής σύστασης προς τα κράτη-μέλη να θαρρύνουν τους φορείς να λάβουν οικονομικές εξασφαλίσεις και ε, εναρμόνισης μέσω ασφάλισης. Ας πούμε στη σύσταση για το shale gas, για το σχιστολιστικό ε, αέριο, ε, αναφέρεται το θέμα μιας οικονομικής εξασφάλισης ή κάποιας αντίστοιχης εξασφάλισης ε, που θα καλύπτει τις ε, διατάξεις της άδεια και τις πιθανές ευθύνες για περιβαλλοντική ε, βλάβη. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην ELD. Το ίδιο γίνεται και για την οδηγία Offshore Safety. Υπάρχουν παρόμοιες διατάξεις. Δυστυχώς υπάρχει αυτός ο κίνδυνος όμως της αφαιρεγγιότητας και πρέπει να σας θυμίσω το Κολοντάρ στην Ουγγαρία 4 Οκτωβρίου του 2010. Εκεί η Ουγγρική κυβέρνηση δαπάνησε σχεδόν 128 εκατομμύρια ευρώ. Για ποιο λόγο, για την αποκατάσταση ε, ενός ε, ε, μιας βλάβης και ο υπεύθυνο μπόρεσε να καλύψει μόνο τα 40.000 ευρώ. Στο Μόρντιξ στι κάτω χώρε, 5 Ιανουαρίου του 2011, οι οικονομικέ εξασφαλίσει δεν ήταν επαρκείς και η τοπική αυτοδιοίκηση πήρε μόνο 50 εκατομμύρια από τα κόστος της αποκατάστασης της βλάβης. Έτσι λοιπόν, αν προκύψει η περιβαλλοντική ζημία, το κόστος της μπορεί να είναι εξαιρετικά μεγάλο. Άρα ο κίνδυνος της αφαιρεγκαιότητας είναι πραγματικός, άρα δεν θα πρέπει να έχουμε ένα ε, καθεστώς αντικειμενικής ευθύνης χωρίς ε, οικονομικές εξασφαλίσεις. Θα υπάρχει ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της οδηγίας σε εκείνες τις περιπτώσεις που ο φορέας ε, δεν θα μπορούσε σε άλλη περίπτωση να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση. Θα διασφαλίσουμε έτσι την ε, αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Ε, ποια είναι τώρα τα εργαλεία ε, οικονομικής εξασφάλισης ή ασφάλεια. Αλλά υπάρχουν και οι τραπεζικές εγγύησεις, αυτασφάλιση, ε, ειδικά ταμεία ε, ή ακόμα και πιο μακριά να πάμε, να περάσουμε μέσα από το επίπεδο το επιχειρηματικό. Εγώ θεωρώ ότι η θεωρία, ε, μάλλον κατανοώ ότι η θεωρία πολλές φορές είναι μακριά από την πράξη και οι εταιρείες στην ουσία θέλουν να παράγουν. Όμως ε, υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του να μην κάνεις τίποτα και το να έχεις οικονομικές εξασφαλίσεις. Μπορεί να υπάρχουν κάποια όρια, μπορεί να υπάρχουν ε, εταιρείε ε, με μικρό κίνδυνο που να έχουν κάποια εξαίρεση, αλλά υπάρχουν πολλές γενικά ευκαιρίες ε, και δυνατότητες που μπορεί κανείς να ε, εξετάσει. Επίσης πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ασφάλιση, γιατί όταν μιλάμε για ασφάλιση, καλύπτει το μισό κίνδυνο, δεν είναι τα πάντα και Υπάρχει και ηθική βλάβη και τέτοια ζητήματα, ηθικός κίνδυνος, κάποιες εξαιρέσεις, ρήτρε κτλ. που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Αν λοιπόν ενσωματώσουμε αυτό το υποχρεωτικό καθεστώς οικονομικών εξασφαλίσεων, θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Για παράδειγμα, ποιοι είναι αυτοί οι φορείς, για ποιο ποσό μιλάμε, ποια είναι τα μέσα που είναι επιλέξιμα, ποια, ποιοι είναι οι όροι κάλυψης που είναι αποδεκτοί και επιτρέπουμε εξαιρέσεις, για παράδειγμα, σε εταιρείε που έχουν εμάς. Τελείωσα μάλλον πιο πριν από ό,τι έπρεπε, οπότε θα έρθω στην, ε, στο συμπέρασμά μου. Όπως είπα και πριν, και το επαναλαμβάνω, η απώλεια της υποχρεωτικής οικονομικής εξασφάλισης δημιουργεί πρόβλημα διότι όταν ένας φορέας θεωρήσει ότι η αντικειμενική ευθύνη για την ζημία ε, που προκύπτει σε επίπεδο ποσών ξεπερνάει τη δυνατότητά του δεν θα πάρει τη βέλτιστη φροντίδα. Θεωρητικά λοιπόν με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσουμε την αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Ας μην έχουμε λοιπόν αντικειμενική ευθύνη χωρίς υποχρεωτική οικονομική εξασφάλιση. Και φυσικά πρέπει να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ κόστους και ωφέλους ε, για την πλήρη ε, προστασία για να έχουμε μια ε, ισορροπία μεταξύ της πλήρους ε, ασυνειδησίας και της αδυναμίας κάλυψης της ευθύνης. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την πολύ ξεκάθαρη παρουσίαση. Ο κύριος Κάμεντα έχει το λόγο. Εκτός μικροφώνου. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις ε, ενδιαφέρουσες και λεπτομεριακή παρουσίαση. Θα δώσω αμέσω το λόγο στον εκπρόσωπο της ε, ομάδας ad hoc ε, που Natural Resources Management Group που προσωπεί τη βιομηχανία καθώς επίσης και τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Διαχειριστών Κινδύνου θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Πιρέντα και μετά τον κύριο ε, Καναμέρας. Ε, σας ζητώ συγγνώμη, έχετε πέντε λεπτά ο καθένας στη διάθεσή του. Κύριος Πιρέντα, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό σα απόγευμα, ε, αξιότιμα μέλη της ε, Επιτροπής. Ονομάζομαι Μάρκο Πιρέντα. Είμαι υπεύθυνο σχέσεων με τις κυβερνήσει, τη ENI. Σήμερα εκπροσωπώ την ομάδα Ad Hoc Industry Natural Resource Management ε, Group, ε, Ad Hoc ομάδα, εργασία, ε, ομάδα της βιομηχανίας. Πρόκειται για μια ομάδα στην οποία συμμετέχουν επιχειρήσεις όπως η ΕΝΑΗ, η ΕΝΑΗ δραστηριοποιείται σε, πολλές, σε πάνω από 16 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τύρο πάνω των 90 δισεκατομμύριων ευρώ. σήμερα δυστυχώς η εκτελεστική διευθύντρια της ομάδα, η κυρία Γκόρντμαν, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω ανηλυμένη υποχρέωση. Εξαιτία και του περιορισμένου χρόνου που έχω στη διάθεσή μα, θα σα αναγνώσω μόνο συγκεκριμένα μέρη ε, τη γραπτή δήλωση που είχαμε προετοιμάσει. Θα σα δώσω πρώτα κάποιε γενικέ πληροφορίε για την ομάδα μα ε, και το πώ έχει δραστηριοποιηθεί στον ε, τομέα τη ε, ε, οδηγία ELD. Θα περάσω μετά σε μια αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα η ELD και κάποιε προτάσει για το πώ μπορούμε να κινηθούμε στο μέλλον. Η ad hoc ομάδα εργασίας ad hoc Industry Natural Resource Management Group δημιουργήθηκε το 1988 και σε αυτήν συμμετέχουν πολυεθνικές ε, εταιρείε και έχει ασχοληθεί με το ζήτημα της αστικής ευθύνη για ζητήματα δικαίου περιβάλλοντος από την αρχή ερχόμαστε σε επαφή με πολλού άλλου φορεί και οργανισμού, όπω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα τη Γενική Διευθύνση Περιβάλλοντο, ε, με εκπροσώπου ε, των επιχειρήσεων, εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών και άλλων. Εμεί θεωρούμε ότι μέχρι στιγμή η ELD λειτουργεί και επιτυγχάνει τους στόχους όμως χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να συλλέξουμε περισσότερες ε, πληροφορίες για συγκεκριμένε υποθέσεις, συγκεκριμένε περιπτώσεις για να αξιολογήσουμε το κατά πόσον ήταν αποτελεσματική. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ίσως υπάρχουν ε, τρόποι να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί χωρίς να ε, μεταβάλουμε το κείμενο της οδηγίας. Η... Η LDE βασίζεται στην πρόληψη και είναι κάτι το οποίο θεωρεί σημαντικό και ο ίδιο ο κλάδο. Βεβαίω, σε συνδυασμό με την ετοιμότητα που πρέπει να υπάρχει σε περίπτωση ατυχήματο. Η LDE συνεχι... Ε, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από πολιετές έργο και έχει ήδη η ομάδα μας συμμετάσχει στην διαμόρφωση αυτής της οδηγίας και έχουμε προγραμματίσει και να συμμετάσχουμε και στην υπόλοιπη ε, συζήτηση όπως περιγράφουμε στη γραπτή μας δήλωση προσπαθούμε να διευκολύνουμε την επικοινωνία και την συνεργασία μεταξύ των, των επιχειρήσεων, του κλάδου ε, και των κυβερνήσεων. Η ομάδα μας θεωρεί και συνεχίζει να θεωρεί ότι η ELD είναι ε, ορθή, είναι κατάλληλη για να επιτύχει τον στόχο της ε, για την προστασία του περιβάλλοντος πέραν της ELD βεβαίως υπάρχει και νομοθεσία των, ε, εθνική νομοθεσία των κρατών μελών και διεθνείς συμβάσεις. Αξιολογώντας λοιπόν όλο αυτό το νομικό πλαίσιο, διαπιστώνουμε ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πεδίο εφαρμογή και την τις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται η ELD. Τις μεγάλες αυτές επιχειρήσεις έχουν εξετάσει τις δικές τους δραστηριότητες για να δουν ε, εάν ε, καλύπτονται αυτές από την ELD. Θεωρούν οι περισσότεροι λοιπόν ε, οικονομικοί επιχειρηματίες σε αυτόν τον τομέα αυτό ότι χρειάζεται να εφαρμοστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήρως η υποχρεωτική ασφάλιση. Και επίσης ότι οι προβλέψεις της ELD σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουν στους παραγωγούς, της δραστηριοποιημένους σε αυτές τις επιχειρήσεις να αποφύγουν την αστική τους ευθύνη. Είχαμε συμφωνήσει και συμφωνούμε μάλλον με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην προτείνει αλλαγές στην ELD αυτή τη στιγμή Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα, χρειάζεται να αποσαφινιστούν έννοιες όπως το, το κατόφλι και ε, χρειάζεται να και θα συνεχίσει μάλλον η ομάδα μας να εργάζεται ώστε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την εφαρμογή της ELD. Ε, έχουμε λάβει γνώση του πολιετούς προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2017-2020 για την ELD, ε, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, έτσι ώστε να ε, λάβουμε και περισσότερες πληροφορίες και ιδιαίτερα πληροφορίες που αφορούν στην υποχρεωτική ασφάλιση. Τι προτάσει μα τι συγκεκριμένε θα τι βρείτε στη γραπτή μα δήλωση, αλλά νομίζω προκύπτει ξεκάθαρα και από τη δήλωση ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακολουθούν ε, και ενδιαφέρονται ενεργά για ε, την εφαρμογή της ELD. Συνεργαζόμαστε με τις εθνικές αρχές. Είναι σημαντικό να μην υπάρχουν στρεβλώσει στον ανταγωνισμό, να είναι ισότιμο ο ανταγωνισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επομένω, οι όποιε αλλαγέ θα πρέπει να ε, εισαχθούν προσεκτικά συνιστούμε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εφαρμογή αυτής της οδηγίας και να μην προβεί αυτή τη στιγμή σε τροποποιήσεις οι οποίες θα ήταν πρόορες ε, και ανέτειες. Θέλουμε να συνεχίσουμε λοιπόν την ε, συνεργασία μαζί σας σε αυτό το πνεύμα και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δώσετε να απευθυνθούμε στην Επιτροπή σας. Σα ευχαριστούμε κύριε Πυρέντα. Ζητώ συγγνώμη που αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε το χρόνο τη παρέμβασή σα τόσο πολύ. Βεβαίω, ε, θα θέλαμε να σα ενημερώσουμε ότι αν θα θέλατε να προσθέσετε στα πρακτικά ε, της ε, Επιτροπής μας τη γραπτή σας δήλωση ε, μπορείτε να τη δώσετε στη γραμματεία και ευχαριστώ θα γίνει αυτό. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Καναμέρα. Ε, πάλι για πέντε λεπτά και πάλι σα ζητώ συγγνώμη. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω την τιμή να α, κάνω αυτή την παρουσίαση ενώπιν της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Γενικός Γραμματέας της ΦΕΡΜΑ, μιας Ένωσης ε, Διαχειριστών Κινδύνων. Και θα ήθελα, θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. εκπροσωπούμε τις εταιρείες διαχείρισης κινδύνου και τις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη που φροντίζουν για την ανάλυση του κινδύνου και την κάλυψή του. Η πρόληψη είναι στην καρδιά του επαγγελματό μας. Και ως εκ τούτου μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου. Θα θέλαμε λοιπόν να συνεισφέρουμε κι εμείς με θετικό τρόπο στην περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να προωθηθούν τα μέτρα πρόληψης για να μειωθεί ο περιβαλλοντικός κίνδυνος. Η ΦΕΡΜΑ συμφωνεί με τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή ότι χρειάζεται να εισαχθούν νέες έννοιες, νέες ε, ρυθμίσεις στην εθνική νομοθεσία έτσι ώστε να εναρμονιστούν ε, σταδιακά οι σχετικές νομοθεσίες, για παράδειγμα όπως συνέβη με την αρχή ο Ριπέν πληρώνει. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ELD. Και θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη των κρατών μελών προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή στην πλήρη αξιοποίηση της ELD, χωρίς να υπάρξουν αυτή τη στιγμή αλλαγές. Ε, ε, έχουν σημειωθεί εξέλιξεις και στον τομέα της αγοράς των ασφαλίστρων κάλυψης περιβαλλοντικού κινδύνου. Με τρόπο ο οποίος να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, αυτό. Ε, η, AIG, η Allianz, μεγάλες επιχειρήσεις του, του κλάδου των ασφαλίσεων έχουν ξεκινήσει να δραστηριοποιούνται και εκεί. Αυτέ οι εξελίξεις είναι θετικέ για όλους και για τις επιχειρήσεις και για την κοινωνία γενικά και για την ε, κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε λοιπόν μέτρα πρόληψης. Με... Ο υπεύθυνο για την αξιολόγηση κινδυνού, ε, αφού ε, αξιολογήσει ποιε είναι οι πιθανές επιπτώσεις ενός ατυχήματος, κάνει κατάλληλες συστάσεις στις επιχειρήσεις. Να σα δώσω ορισμένα παραδείγματα. Ε, σε περιπτώσεις ενός περιβαλλοντικού ατυχήματος ε, και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί για την προστασία της χλωρίδας, της τοπικής ή των ενδυμικών ε, ειδών που μπορούν να ζουν σε ένα, σε ένα οικοσύστημα. Μια άλλη αρχή που προσπαθεί προσπαθούμε να ακολουθήσουμε είναι ότι το ρίσκο θα πρέπει και η επένδυση που θα γίνει για την αντιμετώπιση αυτού του πιθανού ρίσκου, αυτού του πιθανού κινδύνου να είναι η μικρότερη δυνατή. Και άρα χρειάζεται επένδυση στα μέτρα πρόληψης. Η προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί είναι προσαρμοσμένη στην κάθε επιχείρηση. Και βεβαίω η ασφάλιση έναντι του περιβαλλοντικού κινδύνου γίνεται εθελοντική ε, βάση. Η εταιρεία η ασφαλιστική προτείνει προϊόντα τα οποία να είναι προσαρμοσμένα ε, στις πολλές και διαφορετικές ε, δραστηριότητες και είδη επιχειρήσεων που υπάρχουν στην Ευρώπη. Αυτή η διαφορετικότητα θα πρέπει να διασφαλιστεί. Και γι' αυτό το λόγο η Φέρμα ανησυχεί για αυτή την πιθανότητα να εισαχθεί υποχρεωτική ασφάλιση. Γιατί δεν θα αλλάξει τίποτα σε σχέση με τη συχνότητα των ατυχημάτων, ούτε θα αλλάξει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να, επι, να, να επενδύσουν στην ασφάλισή τους εναντί ε, περιβαλλοντικού κινδύνου. Ε, τίθενται ερωτήματα επίσης τεχνικού χαρακτήρα πώς θα προσδιοριστεί ε, με τρόπο που να μην είναι αυθαίρετος το ποσό της, του ασφαλίστου. Και εάν αναγκάσουμε τις επιχειρήσεις ταυτόχρονα να πρέπει να επενδύσουν σε μέτρα πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων, γενικά μέτρα υπέρ τη προστασία του περιβάλλοντο και ταυτόχρονα να αναγκάσουμε να έχουν τέτοιου τύπου ασφαλίσεις, αυτό μπορεί να έχει δεσμενή ε, σε επιπτώσει για την αγωτηγωνιστικότητά του. Είναι δύσκολο ήδη να βρεθεί, να βρει μια επιχείρηση που το επιθυμεί αυτό, μια τέτοια ασφάλιση εξαιτία του μακρόχρονου χαρακτήρα της. Η σταθερότητα ε, είναι ε, απαραίτητος, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ε, για να ασφαλιστεί μια επιχείρηση. Γνωρίζουμε όλοι ότι ένας από τους βασικούς στόχους της ELD ήταν η πρόληψη των περιβαλλοντικών ατυχημάτων και αυτή η η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης δεν πρόκειται να αλλάξει τη συχνότητα των ατυχημάτων. Κατά την άποψή μας, αντιθέτω αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε θα είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στην πρόληψη και στην διαχείριση των κινδύνων. Κλείνω. Θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στην συζήτηση που έχει ανοίξει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα και πιστεύουμε ότι σε αυτό τον διάλογο θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη, στις αρχές της διαχείρισης κινδύνου. Και η πρωτοβουλία για το εφνομοθετήν που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνει τη δυνατότητα να την εφαρμόσουμε στην ELD και αυτό τι σημαίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση ότι η ELD δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί και αν δεν την τροποποιήσει ανέτεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα δώσει ένα θετικό μήνυμα και στον κλάδο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο μιλητές και τώρα συνεχίζουμε τη συζήτηση και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κάσμαν νομικό εμπειρογνώμονα στην Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει το λόγο και να μας εξηγήσει το πολιετές ε, πρόγραμμα εργασίας CRLD που ανέφεραν και οι ομιλητές. Έχετε το λόγο κύριε Κάσμαν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και τις δύο επιτροπές uh, για την ε, πρόσκληση για να σας πούμε κάποια πράγματα για το πολιετές πρόγραμμα εργασίας. Ε, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από το 2017 και θα συνεχίσει μέχρι το 2020 και αποτελεί συνέχεια της ε, έκθεσης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2016 για την εφαρμογή της οδηγίας και η αξιολόγηση που αναφέρθηκε επίσης νωρίτερα σήμερα το απόγευμα. Ε, η αξιολόγηση για το refit μας έδειξε ότι η οδηγία κατά πάσα πιθανότητα επιτυγχάνει πολύ μικρό τμήμα των δυνατοτήτων της ε, για την αποζημίωση και τα ε, αντισταθμιστικά μέτρα για τις ζημίες που προκαλούνται. Θα μπορούσαμε να αναλάβουμε αρκετές δράσεις για να δούμε και να βελτιώσουμε πώς χρησιμοποιείται η οδηγία και αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει τώρα το πρόγραμμα εργασίας. Το πρόγραμμα εργασίας ε, περιλαμβάνει τρεις ε, βασικούς τομείς εργασίας. Ο πρώτος τομέας εργασίας αφορά ε, τις εργασίες βάσει αποδεικτικών στοιχείων, όπως τα αποκαλούμε, πώς εφαρμόζονται στην πράξη λοιπόν κάποια πράγματα στα κράτη-μέλη και θεωρούμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στις πληροφορίες για το πώς εφαρμόζεται η οδηγία. Ένα παράδειγμα αφορά τον αριθμό των περιστατικών και των ατυχημάτων τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν το ένασμα για την εφαρμογή της οδηγίας. Κάποια κράτη-μέλη τηρούν μητρώα αυτών των περιστατικών και ατυχημάτων, αλλά πολλά δεν τηρούν μητρώα και αυτό φυσικά δημιουργεί ερωτηματικά για το ε, πόσες ε, περιπτώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε χρήση της οδηγίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα τέλη του προηγουμένου έτους ε, προσλάβαμε κάποιον εξωτερικό ε, συμβαλόμενο για να μας βοηθήσει να βολτιώσουμε αυτές τις ε, ε, διαδικασίες συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και ένας από τους τρόπους που εφαρμόζεται είναι να εφαρμόζεται ένα σύστημα πληροφορικής για την καταγραφή των πιθανών ε, περιπτώσεων περιβαλλοντικής ευθύνης ε, και αυτές οι περιπτώσεις στη συνέχεια χρησιμοποιούνται, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μάλλον για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή της οδηγίας. Επίσης εξετάζουμε ε, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε μια σειρά ποδίκτες για να δούμε πώς λειτουργεί στην πράξη η οδηγία στα διάφορα κράτη-μέλη και αυτό φυσικά ε, συνάδει και με μια άλλη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, την ε, αναθεώρηση της περιβαλλοντικής εφαρμογής. Εκεί εξετάζουμε με πιο στρατηγικό τρόπο πώς εφαρμόζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία σε κάθε κράτος μέλος και προσπαθούμε να βρούμε βασικούς τομείς στους οποίους θα μπορούσαμε να έχουμε βελτιώσεις. Η πρώτη σειρά εκθέσεων αναχώρα δημοσιεύτηκε νωρίτερα στην αρχή του έτους και ένα από τα θέματα που εξετάσαμε ήταν τα θέματα της οδηγίας της περιβαλλοντικής ευθύνης. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να βελτιώσουμε ε, τις πληροφορίες που δίνουμε εμείς στα κράτη-μέλη για το πώς ε, θεωρούμε ότι λειτουργεί η οδηγία στη χώρα τους και γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη βάση των δικτών που έχουμε για να εξετάσουμε την κάθε χώρα. Ο δεύτερος τομέας εργασίας αφορά το που, καλύπτει το πολιτές πρόγραμμα εργασία, περιλαμβάνει μέτρα τα οποία εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη και αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει μέτρα όπως κατευθυντήριες γραμμές ή προγράμματα κατάρτισης. Έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα για το 2018 και το 2019. Προσπαθούμε στη διάρκεια αυτή της διετίας ε, να προσπαθήσουμε να έχουμε κοινή συνεννόηση για αρκετές έννοιες που αναφέρονται στην οδηγία και άλλοι ομιλητέ ε, σήμερα επεσήμεναν κάποια από τα ερωτηματικά που αφορούν για παράδειγμα την έννοια της περιβαλλοντικής ζημίας, ε, την έννοια της ζημίας στη βιοπικιλότητα που αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα. Ελπίζουμε λοιπόν να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη, με τους εμπειρογνώμονες για να προσπαθήσουμε να ε, έχουμε μια κοινή αντίληψη των ενιών αυτών ε, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να έχουμε καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας. Και εξετάζουμε και άλλες δραστηριότητες ε, στα πλαίσια αυτού του γενικού κλάδου. Ε, τέλος, ένας ακόμα τομέας στον οποίο έχουμε επικεντρωθεί ε, είναι η οικονομική ε, ασφάλεια, η χρηματοοικονομική μάλλον ασφάλεια. Το πρόγραμμα εργασίας αυτή τη στιγμή εξετάζει Ε, project τα οποία αναλαμβάνει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επιθεωρητών ε, για τη χρηματοοικονομική ασφάλεια. Αυτό το έργο ξεκίνησε επειδή υπήρχαν ανησυχίες από αρκετά κράτη-μέλη διότι ο φορολογούμενος ε, στα κράτη-μέλη αυτά στην ουσία ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει για κόστος καθαρισμού, αποζημιώσεις κλπ. σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμα και περιπτώσεις που αφορούν την οδηγία περιβαλλοντικής ευθύνης. Οι εμπειρογνώμονες ε, στην ΙΜΠΕΛ εξετάζουν πρακτικούς τρόπους μέσω των οποίων θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη για να βρουν ποιες είναι οι καλύτερες και πιο αποτελεσματικές ε, μορφές χρηματοοικονομικής ασφάλειας ε, για την κάθε περίπτωση και πώς μπορούμε εν γέννη να βελτιώσουμε την όλη χρηματοοικονομική ασφάλεια σε σχέση και με την οδηγία περιβαλλοντικής ευθύνης αλλά και ε, με μια σειρά άλλα ε, περιβαλλοντικά μέτρα όπως για παράδειγμα αυτά που είναι στον τομέα των αποφλήτων και των βιομηχανικών εκπομπών. Το πρόγραμμα εργασίας μας ε, είναι ε, ένα γενικό πρόγραμμα. Δεν έχουμε καθορίσει τα πάντα για τα επόμενα χρόνια. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν και πώς ε, θα προχωρήσουν η διαδικασία και όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη αλλά και σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένων ε, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων οι οποίοι ήταν εδώ παρόντες σήμερα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και γιατί ήσασταν μέσα στα χρονικά όρια. Άρα έχουμε και τη δυνατότητα για ερωτήσεις ε, προς τους ομιλητές. Έχουμε 20 λεπτά περίπου στη διάθεσή μας για ερωτήσεις και απαντήσεις. Να δώσω το λόγο στους βουλευτές για να θέσουν ερωτήσεις. Δύο, βλέπω. Προτείνω να μαζέψουμε κάποιες ερωτήσεις και από εκεί και πέρα να δώσουμε το λόγο για, ερωτήσεις, για απαντήσεις. Η κυρία Χάουτελα πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήμουν μέλος της Επιτροπής ε, όταν ε, ξεκίνησε η διαδικασία για αυτήν την ε, οδηγία και όταν θεσπίστηκε η οδηγία. Είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να βλέπει κανείς τις ε, επιπτώσεις, τα αποτελέσματα. Αν δεν κάνω λάθος, η Κομισιόν θεωρεί ότι η εφαρμογή θα βελτιωθεί επαρκώς μέσω αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής συμβουλών με τα κράτη-μέλη για καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας. Αν κατάλαβα όμως σωστά, οι ειδικοί μιλούν για νομοθετικές αλλαγές ζητούν τέτοιες αλλαγές. Ίσως λοιπόν θα μπορούσε να αλληλεπεδράσει η Κομισιόν με τους εμπειρογνώμονες και να συζητήσει ενώπιόν μας για την ανάγκη ε, νομοθετικών αλλαγών για τον ορισμό και για, τις, ε, και για τα αμυντικά επιχειρήματα. Νομίζω ο κ. Γκάσμαν ανέφερε αυτό το θέμα, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει ανάγκη να αλλάξουν όλα αυτά να μειωθούν ή να καταργηθούν τελείως ε, οι δύο αυτές, ε, τα δύο αυτά επιχειρήματα λόγω άδειας και λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας. Ευχαριστώ. Οι ομιλητές μπορούν να απαντήσουν γιατί υπήρξαν ε, βέβαια και διαφορετικές απόψεις για συγκεκριμένα ζητήματα. Τώρα, παρακαλώ, έχετε το λόγο για ερώτηση ή σχόλιο. Ε, είμαι ο Πίτερ Τέφερ, είμαι δημοσιογράφος στον EU Observer. Μία από τις περιπτώσεις μέγιστης περιβαλλοντικής ζημίας στο παρελθόν είναι η μόλυνση του αέρα. Και φυσικά οι αυτοκινητοβιομηχανίες που φτιάχνουν δίζελ ε, έχουν μεγάλη ευθύνη γι' αυτό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ELD, ρωτώ την Κομισιόν, για να εφαρμόσουμε αυτή την αρχή του ορυπαίνων πληρώνει στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Ε, βέβαια αυτό το ρωτώ γιατί η ποιότητα του αέρα δεν αποτελεί τμήμα της ELD, του πεδίου της. Θεωρεί η Κομισιόν, οι ομιλητές ε, οι ευρωβουλευτές ότι πρέπει να αλλάξει η ΕΛΤΗ για να συμπεριλάβει την ποιότητα του αέρα για να μπορέσουμε να προλάβουμε τέτοια γεγονότα στο μέλλον. Ευχαριστούμε. Από τη δική μου πλευρά να πω κι εγώ κάτι ως εισηγητής της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να ανοίξει το πεδίο της ELD και να συμπεριληφθεί η ποιότητα του αέρα. Γιατί είναι ένα από τα βασικά μειονεκτήματα της υφιστάμενης οδηγίας. Ε, δεν μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε να, τη σύνδεση αιτίου αιτιατού μεταξύ της αυτοκινητοβιομηχανίας και της μόλυνσης του αέρα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, το κατάλληλο σύστημα ευθύνης για αυτά τα θέματα. Μιλάμε λοιπόν υπέρ της συμπερίληψης της ποιότητας του αέρα και της μόλυνσης του αέρα στο πεδίο εφαρμογής της ELD, αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι και πολύ εύκολο. Βιώνουμε μεγάλη αντίσταση. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο για απαντήσεις δεν ξέρω αν οι ομιλητές, η Κομισιόν, ποιος θέλει να απαντήσει ε, στις ερωτήσεις που έθεσε η Χάιντι Χάουταλα. Δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Is... Ε, μια απάντηση. Ε, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, όπως ο ορισμός της περιβαλλοντικής ζημίας. Είναι πολύ επιστημονικός. Και τα αμυντικά επιχειρήματα, τα οποία προκαλούν δυσαρμονία. Νομίζω φυσικά και κατανοώ ότι υπάρχει πολιτικό πρόβλημα εδώ. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει ένα κείμενο. Η ELD υφίσταται εδώ και 18 χρόνια αλλά η διαδικασία ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια. Υπάρχουν πολλές προτάσεις ε, που κατατέθηκαν και άλλαξαν χιλιάδες φορές και υπήρχε μεγάλη πίεση από τον επιχειρηματικό και βιομηχανικό τομέα ε, που ήταν απέναντι στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αυτά που έχω να πω λοιπόν είναι κοιτάξτε την ιστορία. Αν δεν μπορούμε πολιτικά λοιπόν να αλλάξουμε τα κείμενα, ίσως είναι πιθανό να τα ε, συγχωνεύσουμε με άλλες ε, οδηγίες για να μειωθεί η ζημία η οποία δεν θα είναι περιβαλλοντική αυτή τη φορά αλλά πολιτική. Στην περίπτωση ας πούμε των αμυντικών επιχειρημάτων, ε, εάν δεν θέλουμε να τις καταργήσουμε, θα μπορούσαμε να τις ενσωματώσουμε στην οδηγία των ε, βιομηχανικών εκπομπών του 2008. Γιατί το άρθρο 27 αυτής της οδηγίας είναι αρκετά ευρύ ώστε να συμπεριλαμβάνει αυτού του είδους την ευθύνη. Έτσι, λοιπόν, από αυτή την άποψη είναι δυνατό να πούμε για παράδειγμα ότι ένας παραγωγός που χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ε, βάζει στην αγορά ένα ελληματικό προϊόν, ένα προβληματικό προϊόν και έχει ευθύνη γι' αυτό. Επίσης, ο κίνδυνος ανάπτυξης είναι ένας ε, τρόπος, το Entwicklungsrisiko από την γερμανική νομοθεσία. Τώρα, όσον αφορά στον ορισμό, Συνεχίζω να λέω ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτόν τον ορισμό ως έχει γιατί κανείς ε, δεν καταλαβαίνει. Είναι πολύ επιστημονικός ορισμός. Οι δικαστές όταν εφαρμόζουν την νομοθεσία δεν καταλαβαίνουν τι λέει γιατί είναι δικηγόροι. Εκτός αν έχουν την υποστήριξη επιστημόνων, αλλά δεν είμαστε στις Ηνωμένε Πολιτείες. Τέλος, να πω ότι Όσον αφορά στην ποιότητα του αέρα, η οδηγία δεν το καλύπτει, αλλά αυτό πάντοτε είχε να κάνει με τον ορισμό της περιβαλλοντικής ζημίας, διότι ο ορισμός αυτός δεν λαμβάνει υπόψη τη διαφορά μεταξύ αβιωτικού και βιωτικού. Η οδηγία δεν λαμβάνει υπόψη επίσης την παρέμφαση που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων μέσων, δηλαδή της γης, του αέρα και του νερού. Κοιτάξτε την αμερικανική ε, νομοθεσία της Σούρπλα ή τη σύμβαση του Λουγκάνο που ναι μεν δεν ε, ισχύει αλλά είναι μία από τις πιο προηγμένες νομοθεσίες. Κοιτάξτε πώς έχουν σχεδιάσει αυτό τον ορισμό. Είναι πολύ δύσκολο και είναι και κρίσιμο σε επίπεδο ασφαλίσεων γιατί αν δεν υπάρχει ξεκάθαρος ορισμός για την περιβαλλοντική ζημία πώς θα λειτουργήσει ο ασφαλιστικός ε, κλάδος, πώς θα ποσοτικοποιήσουμε την περιβαλλοντική ζημία. Και το, θέλω, το θέμα δεν τελειώνει εδώ. Τι γίνεται με τις εκπομπές, ε, με τις ζημιές ε, στις οποίες δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τη σχεση εντοπίσουμε το φορέα, τι γίνεται. Είναι περίπλοκα τα αιτίο-αιτία του ή όταν δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τον φορέα, τι γίνεται. Είναι περίπλοκα τα ζητήματα, χρειάζεται μία ισορροπία μεταξύ των διαφόρων κλάδων. Η βιομηχανία δεν μπορεί να τα έχει όλα δικά της, κάτι πρέπει να γίνει. Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο, αρχίστε να ε, συγχωνεύετε με άλλες ε, οδηγίες. Ευχαριστώ. Κάποια άλλη αντίδραση να θέσω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις απευθείας στους ομιλητές. Η μία ερώτηση είναι για τον κύριο Γκερέντα και τον κύριο Καναμεράς. Και οι δύο αναφέρατε ότι σύμφωνα με την εμπειρία σας οι βιομηχανικές εταιρείες θεωρούν ότι δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω νομοθεσία και ρύθμιση και ότι δεν χρειάζεται κάποιο υποχρεωτικό σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας, ότι υφίσταται στην ELD αρκεί. Ε, η ερώτησή μου προς τους δυο σας είναι κάτι που δεν θα σας εκπλήξει φυσικά. Συνήθως οι εταιρείες και επιχειρήσεις δεν ενθουσιάζονται με τη μεγαλύτερη ρύθμιση και τις περισσότερες νομοθεσίες, όμως αυτό που έχουμε στην Ευρώπη με την ELD είναι ε, μια προχειροδουλειά που ε, συνενώνει διαφορετικά οικονομικά και ασφαλιστικά συστήματα. Σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν συστήματα περιβαλλοντικής ασφάλειας, αλλά όχι. Αυτό δεν είναι ίσοι σε κάποια τμήματα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς υπάρχουν διαφορετικοί όροι για τις εταιρείε από τις άλλες. Κάποιες ε, χώρες λοιπόν είναι πιο φθηνές, οπότε κανείς ε, μπορεί να ρηπαίνει χωρίς να δαπανά χρήματα γιατί δεν υπάρχουν υποχρεωτικές ας πούμε εξασφαλίσεις. Υπάρχουν επίσης και προβλήματα με την ε, νομοθεσία για τον ανταγωνισμό κατά τη γνώμη μου. Καταλαβαίνω λοιπόν αυτό που λέτε, αλλά προσπαθώ να πω ότι αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι στην ουσία μια εναρμόνιση της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε λίγη, κάποια περισσότερη ρύθμιση σε κάποια κράτη-μέλη υπό τη σκέπη της ELD για να έχουμε ένα σωστό πεδίο, ίσους όρους, ε, γιατί σε κάποια κράτη-μέλη έχουμε διαφορετικά καθεστώτα περιβαλλοντικής ευθύνης από άλλες. Ε, θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια εναρμονισμένη προσέγγιση κατά τη γνώμη σας. Και η δεύτερη ερώτηση στον κύριο Κάσμαν. Αναφέρατε ότι στο πολιετές πρόγραμμα εργασίας της η Κομισιόν κυρίως επικεντρώνεται στην καλύτερη εφαρμογή της ELD, δεν την ανανεώνει, δεν ξανανοίγει τη συζήτηση για επιπλέον νομοθετικές δράσεις. Νομίζετε όμως ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία τα βιώνει ήδη η Κομισιόν. Για παράδειγμα, όταν έγινε η μελέτη εφαρμογής για την ELD, είδαμε ότι τα κράτη-μέλη κατανοούν την οδηγία με τελείως διαφορετικό τρόπο. Απλά πράγματα, όπως ο τρόπος που αναφέρουν στοιχεία στην Κομισιόν. Διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Το 75% των αναφορών είναι από δύο κράτη-μέλη και τα υπόλοιπα δίνουν το υπόλοιπο ποσοστό. Άρα, ε, ίσως καλύτερη εφαρμογή ε, της υφιστάμενης ε, οδηγίας ε, θα μπορούσε να λύσει όλα τα προβλήματα που βιώσατε ή χρειάζεται μία βελτίωση της ίδιας της οδηγίας. Κυρία Φεράρα έχει μια ερώτηση και μετά μπορούμε να επανέλθουμε στις απαντήσεις. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ τους εισηγητές που πήραν τον λόγο. Εγώ είμαι εισηγήτρια μαζί με τον συνάδελφο Γιάβορ για την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για την εφαρμογή της οδηγίας ELT. Θα ήθελα να ζητήσω κάποιες διευκρινήσεις και την άποψή σας, ε, συνδέοντας και τα όσα είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως με το θέμα αυτό. Η διαφορά που αφορά την νομοθεσία σε όλα τα κράτη-μέλη. Σήμερα έχουμε την οδηγία και κατά την άποψή σας πιστεύετε ότι θα πρέπει να ξαναδούμε ε, τη νομική βάση και να γίνει κανονισμός ή μάλλον το νομικό μέσο και να γίνει κανονισμός διότι από τις διάφορες συζητήσεις που έγιναν αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανισότητα μεταξύ των κρατών μελών και μια δυσκολία ε, αντίληψης των πληροφοριών, να έχουμε και κάποιες ε, πληροφορίες και κάποιες αντικειμενικές βάσεις επί των οποίων από εκεί και πέρα θα ε, ε, δούμε λίγο κατά πόσον, πότε και πώς να παρέμβουμε. Το να υπάρχει λοιπόν ένα νομοθετικό μέσο το οποίο να είναι αντίστοιχο για όλα τα κράτη-μέλη, κατά την άποψή μου θα βοηθούσε να υπάρχει εναρμόνιση, να υπάρχει ισότητα δηλαδή, ε, νομικών ε, τάξεων, ένομων τάξεων και αυτό σημαίνει και δυνατότητα να παρακολουθούμε τις διάφορες καταστάσεις στα κράτη-μέλη. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα αφορά αυτό. Μετά, όσον αφορά την παρακολούθηση. Η παρακολούθηση μέχρι τώρα δεν είχε αποτέλεσμα και δεν είχε αποτέλεσμα διότι ε, υπησέρχονται πληθώρα λόγων ε, και λόγω έλλειψης ανεξαρτησίας σε κάποιες περιπτώσεις ε, ε, και των ίδιων των επιθεωρητών, αλλά και γιατί υπήρχαν διαδομένες στα κράτη-μέλη κάποιες δραστηριότητες πριν essere delle attività eh, επιχειρήσεων που ε, κάνουν επικίνδυνες δραστηριότητες για το περιβάλλον. Επομένως και εδώ η ιδέα θα μπορούσε να είναι να έχουμε ένα μητρό, ώστε όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν κάποιες δραστηριότητες, οι οποίες ε, δυνητικά θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά σε αυτό το μητρό, να γίνεται καταχώρηση εκεί και να υπάρχει ε, και διευκόλυνση για τους επιθεωρητές οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν και μια πιο μόνιμη παρακολούθηση. Για τα όσα αφορούν τη χρηματοοικονομική ασφάλιση. Εγώ εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Καναμέρας ως προς το γεγονός ότι η υποχρεωτική χρηματοοικονομική ασφάλιση δεν ε, αντισταθμίζει την περίπτωση περιβαλλοντικού κινδύνου. Δεν ε, αποτελεί αυτή σαν ασταλτικό παράγοντα και καλύτερο θα ήταν ε, να υποστηρίξουμε την πρόληψη και την προώθηση της διαχείρισης του κινδύνου. Έχω πιστεί επ' αυτού, διότι μας το αποδεικνύουν και τα γεγονότα. Εγώ είμαι Ιταλίδα. Ε, είμαι από την Καλαβρία, είμαι από μια περιοχή δηλαδή στην οποία ζούμε με τοξικά απόβλητα ε, και δυσκολευόμαστε ε, να κατανοήσουμε και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα εδάφια αυτά. Ο κίνδυνος δεν είναι μόνο ε, περιβαλλοντικά, υπάρχει κίνδυνος και για τους πολίτες που ζουν εκεί. Υπάρχει όλο ένα αυξανόμενος <laughs> κίνδυνος ε, για την εμφάνιση νεοπλασιών και όγκων ε, λόγω της τοξικότητας της περιοχής. Επομένως θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει και πρόληψη, διότι μετά ε, είναι πάρα πολύ αργά για να επενορθώσουμε μια κατάσταση που μπορεί να χρειάζεται πολύ χρόνο για να επανέλθει στην κατάσταση πριν από την ε, περιβαλλοντική ζημιά. Σίγουρα λοιπόν πρέπει να επικεντρωθούμε στην πρόληψη και στη διαχείριση του κινδύνου, αλλά η αλήθεια είναι ότι μια χρηματοοικονομική ασφάλιση και μια κάποια μορφή οικονομική εγγύηση πρέπει να υπάρχει, διότι δυστυχώ υπάρχουν και επικίνδυνε καταστάσει. Και πολύ συχνά συμβαίνει οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι οι υπεύθυνε να χρεοκοπούν, να εξαφανίζονται και μετά να μην υπάρχει κανένας ο οποίος ε, θα ε, αποζημιώσει και θα αναλάβει το κόστος ε, για την επισκευή της ζημίας ή την επανόρθωση της ζημίας. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν εγγύησει σίγουρα και η διάρκεια έχει μεγάλη σημασία, αλλά πρέπει να βασίζονται και στη δραστηριότητα της επιχείρησης και με βάση αυτά να γίνεται και εκτίμηση της ε, ε, χρηματοοικονομικής ασφάλισης που θα πρέπει να καταβάλει κάθε επιχείρηση. Η εναλλακτική λύση θα ήταν να υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο, αλλά το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, ε, έχει αρκετά θέματα. Ποιος θα τα χρηματοδοτεί, οι πολίτες ε, θα αναλαμβάνουν τη δαπάνη για τη χρηματοδότηση αυτού του ταμείου. έχω κάποιες αμφιβολίες επ' αυτού. Και μια τελευταία ερώτηση που αφορά το θέμα της ε, δευτερογενείους ευθύνης ε, τρίτων ε, που προέρχεται από την ζημία. Πρόκειται για ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο δεν περιλαμβάνεται σήμερα στην οδηγία ELD, υπάρχει όμως σε κάποια κράτη-μέλη και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας την άποψη για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much and now I would give the floor for... Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους ομιλητές μας για να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις, όπως το επιθυμεί. Θα μιλήσω Ιταλικά, εάν δεν έχετε αντίρρηση. Χωρίς μικρόφωνο. As όπως βλέπετε και όπως διαπιστώνετε και από τις ερωτήσεις που ετέθησαν εδώ, οι τεχνικές ε, σκοπιές είναι αυτές οι οποίες μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Με όλο το σεβασμό, επειδή βρισκόμαστε στο μέγιστο πολιτικό οικοδόμημα, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε εδώ πέρα τις ε, δυσκολίες που υπάρχουν σε τεχνικό νομικό επίπεδο. Πρόκειται για οδηγία πλαίσιο, ακριβώς γιατί υπήρχε νομοθεσία δεσπόζουσα και ακόμα έχουν ε, δεσπόζουσα θέση στην ε, ε, εθνική νομοθεσία και επομένω είναι πολύ δύσκολο να το συνδυάσουμε με το ευρωπαϊκό δίκαιο αυτό. Υπάρχουν και παρεμπίπτοντα θέματα, όπως ποινικό δίκαιο, ε, αστική ευθύνη και πολύ διαφορετικό αστικό δίκαιο μεταξύ των κρατών μελών. Επομένως, καταρχήν ε, η απάντηση ε, της κυρίας Φεράρα είναι ότι εμεί είμαστε πάντα υπέρ τη μέγιστη συναρμόνιση. επομένω σε έναν ιδανικό κόσμο ο κανονισμό θα μπορούσε να μα κάνει και ευτυχισμένου, διότι θα υπήρχαν σαφεί κανόνε και δεν θα έπρεπε να πηγαίνουμε στα διάφορα βήματα για να βρούμε τι δίκαιο ισχύει. Αλλά όσον αφορά την τεχνική νομική πρόκληση, ε, για σήμερα θεωρώ ότι είναι αδύνατο, λαμβάνοντα υπόψη το γενικότερο νομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μα. Κάποιε παρατηρήσει πολύ σύντομε για αυτά τα οποία ακούστηκαν για τη συμμετρία στα διάφορα κράτη-μέλη και διάφορες άλλες πτυχές όπως για παράδειγμα το κόστος για τους πολίτες, ε, τους φορολογουμένους ε, για την ε, υποστήριξη του περιβαλλοντικής δαπάνης. Ε, ασφαλιστικές εισφορές και χρηματοοικονομική ασφάλεια. Πολύ μεγάλο κόστος της χώρας μου τουλάχιστον για τους πολίτες δεν αφορά και ελπίζουμε ότι δεν θα αφορά ποτέ στο μέλλον τη ρήπανση ε, μετά από την οδηγία. Αλλά για την περίπτωση στην οποία αναφέρθηκε και η κυρία Βουλευτής αφορά ιστορική ρήπανση. Μπορούμε να σκεφτούμε για παράδειγμα ότι θα υπάρχει ασφαλιστική εταιρεία που θα καλύψει ιστορική ρήπανση για μια ε, περιοχή, για ένα μνημείο το οποίο είναι ορφανό, δεν έχει κάποιο κάτοχο για να σας εξηγήσω και λίγο πόσες τεχνικές δυσκολίες υπάρχουν. Τώρα, όσον αφορά τις εξαιρέσεις, ε, πρόκειται για περιπτώσεις που είναι ε, αυστηρή ερμηνεία της οδηγίας. Για παράδειγμα, στην Ιταλία οι δεύτερες περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται. Ε, δεύτερον, υπάρχουν και κάποιες παράπλευρες συνέπειες τις οποίες δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. Για παράδειγμα, ποινικά θέματα. Μπορεί η επιχείρηση να μην έχει κανένα συμφέρον να χρησιμοποιήσει την, ε, το αμυντικό επιχείρημα της άδεια ε, για την περιβαλλοντική ζημία, αλλά μπορεί ο διαχειριστής της εταιρεία ε, να πρέπει να αποδείξει ότι όσοι είχαν γίνει έγιναν κατόπιν άδεια σε ποινικό επίπεδο. δηλαδή, θα ήθελα να ζητήσω από τους παρισταμένους να προσέξουν πάρα πολύ το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν και τεχνικές και νομικές συνέπειες για την όλη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ ευχαριστούμε. Κύριος Καναμέρας. Θα συνεχίσω στα γαλλικά εγώ. Όπως και στην παρέμβασή μου. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που μόλι υπόθηκε. Πράγματι είναι πολύ περίπλοκη η εναρμόνιση, παρόλο που είναι επιθυμητή από όλους και ιδιαίτερα από τι επιχειρήσεις, γιατί διευκολύνει τη δραστηριοποίησή τους. Όμως, η συνθήκες είναι διαφορετικές από τη μία χώρα στην άλλη. Για παράδειγμα, στην Γαλλία έχουμε ένα δίκαιο για, την, για το περιβάλλον, για την περιβαλλοντική ευθύνη, ήδη προηγμένο και εύκολα ενσωματώθηκε η ΕΛΔΗ. Η εναρμόνιση λοιπόν δημιουργεί προβλήματα, αλλά πίσω από αυτά τα προβλήματα ίσως να είναι τελικά η, η πολιτική συζήτηση που πρέπει να γίνει. Τώρα όσον αφορά την υποχρεωτική ασφάλιση, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε το, ζήτημα το πιο ε, βασικό, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αγορά. Όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής, σε ορισμένες χώρες έχει εφαρμοστεί υποχρεωτική ασφάλιση για την, α, ε, τις περιπτώσεις ρήπανσης του εδάφους ε, και την αντιμετώπιση τους μετά από μια εκμετάλλευση. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει συμφωνία σε αυτά τα θέματα. Για παράδειγμα, είναι, γιατί θα χρειαστεί να συμφωνηθεί το ζήτημα της διάρκειας, του ποσού. Ε, η, μια τράπεζα δεν πρόκειται να δεχθεί μια τέτοια ασφάλιση ε, SAE με απεριόριστη χρονική διάρκεια και θα είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί ακόμα και μια 20 ετή, για παράδειγμα, ασφάλιση. Ε, ιδιαίτερα ε, δεδομένη της κατάστασης του χρηματοοικονομικού συστήματος σήμερα. Βεβαίως, μπορεί κανείς να αξιοποιήσει τι ασφαλιστικέ εταιρείε, αλλά και πάλι θα πρέπει να είναι σαφώ καθορισμένο ο κίνδυνο έτσι ώστε να ποσοτικοποιηθεί και να είναι συγκεκριμένο και το, το, το ποσό της ασφάλισης. πρόβλημα λοιπόν της ισοτιμίας και της ε, εναρμόνισης δεν πρόκειται να λυθεί με τον καταστή ασφάλιση υποχρεωτική. Αντιθέτως θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερη ανισότητα και, ανισορο... Ε, και ε, διαφορές μεταξύ των επιχειρήσεων. θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από το ζήτημα των αποζημιώσεων. Τουλάχιστον να υπάρξει μια συμφωνία σε αυτό ε, και μετά ας προχωρήσουμε στα παραπέρα βήματα βλέποντας και την εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα και στον κύριο Κάσμαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους που ήθελαν να λάβουν το λόγο. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δίνω τον λόγο στον πρόσωπο της Επιτροπής και μετά στον κύριο Καβαντά. Κύριος Κάσμαν για να απαντήσω στο ερώτημα που μου ετέθη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αισιόδοξη όταν υιοθετεί πολυετή προγράμματα εργασίας γιατί θεωρεί ότι υιοθετώντα αυτά τα προγράμματα μπορούμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή της οδηγίας. Όμως, δεν θα αποκλείσουμε το ενδεχόμενο κάποια στιγμή στο μέλλον να θεωρήσουμε, να αποφασίσουμε ότι θα ήταν χρήσιμο να προτείνουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποιήσεις στην οδηγία. Δεν μπορώ να το αποκλείσω λοιπόν. Ωστόσο λέω ότι το πολιτές πρόγραμμα εργασιών συμπεριλαμβάνει και δράσει για την βελτίωση των, της, των στατιστικών στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μα, έτσι ώστε να γνωρίζουμε πώς έχει εφαρμοστεί στην πράξη η οδηγία, έτσι ώστε και σε λίγα χρόνια να έχουμε τη δυνατότητα να ξαναξιολογήσουμε την κατάσταση και να δούμε πού βρισκόμαστε. Δεν θα σας πω λοιπόν ότι ποτέ δεν πρόκειται να προτείνουμε αλλαγές στην οδηγία. Απαντώ επίσης σε μια σειρά ζητημάτων που έθεσε η κυρία Φερέρα. Έχετε δίκιο που τονίσατε την σημασία της πρόληψης. Και εδώ συμφωνώ και με πολλούς άλλους ε, ομιλητές. Η οδηγία ELD δεν θα πρέπει να την βλέπουμε ξεχωριστά ε, ως απομονωμένο νομικό μέσο, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα ε, νομικά εργαλεία για την πρόληψη των περιβαλλοντικών ζημιών. Αν δούμε το παράρτημα 3, που περιγράφεται σε ποιες επιχειρήσεις εφαρμόζεται η αρχή της αντικειμενικής ευθύνης. Πρόκειται για επιχειρήσεις στις οποίες έτσι και εφαρμόζονται και οι προβλέψεις της οδηγίας για τους βιομηχανικούς ρήπους, που είναι πολύ λεπτομεριακές, άρα υπάρχουν και άλλα νομικά εργαλεία για την πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων. Και θεωρούμε ότι είναι πράγματι σημαντικό να συνδέεται η εφαρμογή της ELD με την εφαρμογή αυτών των άλλων νομικών εργαλείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει, έχει προγραμματίσει μάλλον να αναλάβει μια πρωτοβουλία, μια ανακοίνωση για το, τη, γενικότερη, το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο για το περιβάλλον, έτσι ώστε να υπάρξει συνδυασμός της CLD με τα υπόλοιπα νομοθετικά, νομικά εργαλεία έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτά τα πτυχήματα που όλοι θέλουμε να αποφεύγουμε, αυτές τις καταστάσεις που όλοι θέλουμε να αποφεύγουμε και να είναι ξεκάθαρο πώς ανταποκρινόμαστε σε τέτοιου τύπου περιβαλλοντικά συμβάντα εάν συμβούν. Θεωρούμε επίσης ότι αυτό το νομικό πλαίσιο λειτουργεί και αποτρεπτικά Ελπίζω να σας έδωσα ε, κάποιες, μια καλή περιγραφή του πώς βλέπουμε εμεί τα πράγματα και αυτό να σας βοηθήσει τη συζήτησή σας. Ο κύριος Καπαντά. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην εισηγήτρια μα την κυρία Φεραρά, για να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που πήραν το λόγο για τα εξαιρετικά ε, θέματα τα οποία έθιξαν σήμερα, τροφή για σκέψη, σίγουρα είναι σύνθετα αυτά που πρέπει να κάνουμε. Συμφωνώ ότι αφενός πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση μεταξύ όλων των κρατών μελών ε, η οποία θα διευκολύνει λίγο τη ζωή όλων, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την υπόλοιπη νομοθεσία που υπάρχει επί του θέματος. Σαφώς και θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση, όχι μόνο μεταξύ κρατών μελών, αλλά και με την υπόλοιπη σχετική νομοθεσία και να υπάρχουν συνδυασμένες διατάξεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να έχουμε ένα ομογενές πλαίσιο σε θέματα πρόληψης και επανόρθωσης της ζημίας σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Τώρα, όσον αφορά την ιστορική ρήπανση, για να απαντήσω στον κύριο Πυρέντα, ε, πρόκειται για ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε και πιστεύω ότι η νομοθεσία η οποία θα πρέπει να επαναθεωρηθεί δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ. Επομένως, ε, πρόκειται για κάτι το οποίο θα πρέπει να ε, απαντηθεί με άλλο τρόπο. Μελλοντικά όμως ε, σίγουρα θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια νέα στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να μην έχουμε και πάλι ε, συσσόρευση, ρήπανσης ε, και ζημία για το περιβάλλον όπως έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με τον συνάδελφο Γιάβορ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα πρέπει να ξαναδούμε και το κατόφλι ε, και να δούμε και τις δυνατότητες παρακολούθησης και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Στενή ε, επαφή με την Επιτροπή ΕΜΒΗ. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ όλους. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαμε εξηγήσει και ερωτήσει, ε, μπορέσαμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και το οποίο φυσικά θα έχει διάρκεια και στο έργο του νομοθέτη και των ε, νομικών και των τεχνικών και όλων εκείνων που ε, τους ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα, κυρίως των επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και την πειθαρχία σας για να μπορέσουμε να έχουμε μια αποτελεσματική ακρόαση και τώρα θα συνεχίσουμε και κλεισμένο των θερών. Επομένως, εκείνοι οι οποίοι δεν πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα, σας παρακαλώ να αποχωρήσετε από την αίθουσα γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει λίγο και έχουμε αρκετά θέματα στην ημερήσια ε, ε, διάταξη. Ευχαριστώ πολύ και ο πρόεδρος Βόμποντα φαντάζομαι θα αναλάβει και πάλι τα ενία.